Καλό μεσημέρι απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συνήθιστη ώρα για ψηφοφορίες, αλλά παρακαλώ καθίστε. Ξεκινούμε με την πρώτη έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Ονομαστικά θα ψηφίσουμε συνολικά την απόφαση την απαλλαγή άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δεν έχετε ψηφίσει ακόμη όλοι. Jetzt είμαστε 560. 560. Άλλα ακόμη μερικά δευτερόλεπτα ανοιχτή η ψηφοφορία για να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάσαμε γύρω στους 600 τώρα. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 14 ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται τροπολογία 1 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 83 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 85 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 120 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψηφιπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 143, τροπολογία 5 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε, αν και νομίζω ότι απορρίπτεται, άρχεται ψηφοφορία, πρώτο τμήμα της τροπολογίας 5. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πράγματα απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. ψηφίπε. Α, καταπίπτω δεύτερο. Πάμε στο πόγιο εξπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 27. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Την 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται. Συγγνώμη. Η τροπολογία 7. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται το 28 και κυκλήση. άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται τροπολογία 10 ψήφι περ. κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 Α, ελέγχουμε τη 10. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Απολογία 11 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αλλά παρακαλώ να σκόνετε καλά τα χέρια. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ της 8. Κατά. Αποχές. Green Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 17 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 ψήφι υπέρ. Ελέγχουμε την 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε τροπολογία 18 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 ψήφι υπέρ 19 περ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτε τροπολογία 20 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 ψήφι υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται τρόπο 29 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη δεύτερη έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντε. Κυρία Μπερές, έτοιμα της διαδικασίας. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λάβατε αιτήματα ως προς το παράδειγμα ορισμένων διατάξεων. Αρνηθήκατε να λάβετε θέση. Όμως ξεφνικά και κατ' βλέπουμε τον κύριο Βέμπερ, ότι έχουμε εδώ τροπολογίες διαγραφή. Αυτό δεν έχει σχέση με ένα πολιτικό πρόβλημα. Είναι θέμα συνεργασία μεταξύ των επιτροπών. Το περιεχόμενο αυτών των παραγράφων αφορά κρίσεις όσον αφορά το Ταμείο εξηγένση ε, Τραπεζών. Και αυτό δεν είναι, αυτά τα όργανα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Προσέξτε λοιπόν, ε, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές έχουν συνυπογράψει λοιπόν προτάσεις τροπολογιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο τροπολογιών, στον κατάλογο ψηφορίας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητή συνάδελφε, κυρία Μπερέσα, Δεν ε, υπήρξε όμως κάποιο αίτημα για να κυριχθούν οι παραδεκτές κάποιες ε, τόπες. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε στην ένα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνω. Την ένα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Αλλά μπρος και πίσω ε, βλέπω να πηγαίνετε και οχι δεν ξέρει να ψηφίζετε. Λοιπόν, δύο ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Πέντε ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε την πέντε. άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Die Abstimmung Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Άργησα Δυστυχώ να το ακούσω, Κάποιο το φώναξε, αλλά τέλο πάντων. Και τον, για, το, για την 4 έχει ζητηθεί ηλεκτρονικό έλεγχο. ψηφίζουμε. Για την 4 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίθηκε 4. Πηγαίνουμε στην 6 ψήφι υπέρ. Συγγνώμη. Δεν μου είπε κανένα να ψηφίσουμε την 3. Το 4 ναι. Πράγματι κάποιο φώναξε για την πέντε ψηφίσαμε. Ε, δεν είναι ότι πήδησα μία. Ε, λοιπόν, πάμε στην έξι τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την ψηφία, 8 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 ψήφι περ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, την 11 ελέγχουμε με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 12 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το πρωί 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνει τροπολογία 14 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνει τροπολογία 15 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 16 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται 17 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται 18 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Θέλετε να ελέγξουμε το 18, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 ψηφιπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 20 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 ψήφι υπέρ. Ελέγχουμε την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. τρόπο 23 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τρόπο 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος τώρα, όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή η έκθεση. Και πηγαίνουμε στην έκθεση βάλει Αρχικά ψηφίζουμε την απόφαση την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Την τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ναι, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. Ο κ. Τραπέλα, νομίζω, όταν του ζητήθηκε να σηκώσει το χέρι του για την προηγούμενη έκθεση, Αγιάλα Σεντέρ, δεν κατάλαβα τι ψήφισε, γιατί ψήφισε και υπέρ και κατά. Κύριε Πρόεδρε, πώς κάνατε την καταμέτρηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν το έχει κάνει αυτό ο κύριο Ταραμπέλα. Ε, συγγνώμη κύριε Ταραμπέλα, εγώ μιλάω τώρα. <laughs> Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αν Πράγματι το έκανε. Γιατί δεν το, δεν το είδα εγώ προσωπικά. Ακριβώς πρόεδρε, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη δουλειά μας. Εδώ έχω ένα κατάλογο με τροπολογίες ΕΛΚ ε, και σοσιαλιστών. Έλεγε κατά. Ε, και έτσι η δεξιά πλευρά είπε υπέρ, η άλλη κατά. Τώρα δεν νομίζω ότι αυτό μειώνει την ικανότητα του Πρόεδρου να μετράει αν τελικώ το Κοινοβούλιο αυτό είναι υπέρ ή κατά. Θα σας επιτρέψω άλλη μια φορά να πάρετε το λόγο, τη συνάδελφοι, αρκεί να είναι για τη διαδικασία. Ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε εδώ θεατές, έχουμε δημοσιογράφους για τον κύριο Ταμπραμπέλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώς είναι ένα μεγάλο αστείο. Χώρος έκφραση χιούμορ. Ευχαριστώ για την βαθιστόχαστη αυτή παρατήρηση. Πηγαίνουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σμίτα. Καταρχάς, ψηφίσουμε την απόφαση για την απαλλαγή. Ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Ναι, η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 14 σε δύο τμήματα. Το πρώτο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση και αυτό. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, με διορθώνουν ε, την τροπολογία 2 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα που λέει 34. Θέλετε να ελέγξουμε. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 36. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, δύο τμήματα. Ονομαστικά και τα δύο. Πρώτο τμήμα άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, μονομαστική και αυτό ψηφοφορία, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, λοιπόν, το έχουμε ρυθμίσει. Πηγαίνουμε στο αρχικό κείμενο της 40, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 41, αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 42 αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 43. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παράγραφου 44 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 48. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε τμήματα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία του πρώτου τμήματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε το πρώτο Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά πάντα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 36 τροπολογία, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 56 παράγραφος. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολέ 37 μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολέ 32 μονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Προπολογία 17, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προπολογία 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46, ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 80 αρχικό κείμενο. Σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Το προϊόν Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 85. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται 88 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται 91 Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την παράγραφο 88, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράφωση 91 ευκό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 τροπολογία υπέρ. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα του 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 33. Τροπολογία ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το πρωί 38 υπέρ, κατά, εποχέ, απορρίπτεται. Ροπολογία 4, μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 31. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερω αν από την αριστερά τα ε, ψήφιζαν ε, καλά, ε, με σηκωμένα καλά τα χέρια οι συνάδελφοι, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο. Παράγραφος 107 σε 4 με τα πρώτα τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα. Ελέγχουμε. Δεύτερο τμήμα της 107 έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, τρία τμήματα ονομαστικά ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 6. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 7, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφισάτε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 τροπολογία ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στην 109 ε, πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 109 ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παρά 110 αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 ψήφι υπέρ. Κατά. Χμ. Αποχές. Ελέγχουμε. 112 ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 113 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 ψήφι περ. Θέλετε να επαληθεύσουμε τα 113, έχετε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 115 ψήφι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 ψήφι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 ψήφι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ τη 12 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 13 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 39 τώρα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα, κατά πίπτη 27, τροπολογία 21, ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Όπως είπα, κατά πίπτη 27 πηγαίνουμε στην 28. Ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 ψήφι περ, να ελέγξουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Μονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε τώρα στις πολυάρθμες εκθέσεις του κυρίου Κον. Αρντ Κον. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταρχάς για το σύνολο της απόφασης για την αναβολή απαλλαγής υπερκατάποχες εγκρίνεται. Το ψήφισμα συνολικά ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται τώρα έκθεση για το δικαστήριο. Απόφαση για την απαλλαγή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται τώρα έκταση εικόν για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχικά την απόφαση για την απαλλαγή ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται και το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται έκθεση τώρα για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τώρα έχουμε τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 9 σε ιδιωτήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο του με μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση εικόν τώρα για την Επιτροπή των Περιφερειών. Στην απόφαση για την ε, υπερκαταποχέ εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τώρα, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ άπορη. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά Αποχές από τροπολογία ένα, με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση εικόνων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Απόφαση για την απαλλαγή υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 από το ψήφισμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 32. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται το σύλλογο του ψηφίσματο ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση εικόνη για τον Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Για το ψήφισμα τροπολογία 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται και το σύνολο του ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. αφού πρώτα όμως απαληθεύσουμε την ένα ηλεκτρονικά. Ψήσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα Έκθεση για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, απόφαση για την απαλλαγή ψηφιπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται, σύνολο ψηφίσματο. ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε με τον κύριο Κον και πάμε στην άλλη σειρά εκθέσεων του Πέτρη Σαρβάμα. Καταρχά, επιδόσει δημοσιονομική διαχείριση έλεγχου των οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τη 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 σε δύο τμήματα ονομαστικά. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρασε. δεκτό δεύτερο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Αρβάμα για τον ορισμό συνεργασία των εθνιστικών αρχών ενέργεια. Ψήφισμα βλάγει υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ψήφισμα συνολικά. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα η έκθεση Αρβάμα για την υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Θεσμικών Αρχών για τι Εκτονικέ Ποινίε, απόφαση για την απαλλαγή ψηφί υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματο σε ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκτε Αρβαμά για το μεταφραστικό κέντρο των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση την απαλλαγή. Ψηφί Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τώρα έχουμε το αρχικό κείμενο του 18 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος. Μοναστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται τώρα έκθεση Αρβαμά για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματική Κατάρτιση. Απόφαση να μιλάγει υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, σύνολο ψηφίσματος, μονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Αρβαμά για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στο τομέα τη επιβολής του νόμου. Απόφαση για την απαλλαγή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο του ψηφίσματος μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια τη Αεροπορία. Απόφαση την απαλλαγή ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματο ε, με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Αρβαμά τώρα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο. Απόφαση αναβολή απαλλαγή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Αρβαμά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, απόφαση την απαλλαγή ψήφι Κατά αποχέ εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα πηγαίνουμε στην αρβάμα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Αρχικά απόφαση για την απαλλαγή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τώρα σύνολο ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται και τώρα έχουμε την έκθεση Αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Απόφαση την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα έχουμε ε, το αρχικό κείμενο παραγράφου 5. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τι θέλετε να ελέγξουμε την παράγραφο 5 το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε απορρίφθηκε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε εκτεσαρπάμα αρπαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος απόφαση για την απαλλαγή ψήφι Κατά Αποχέ. εγκρίνεται σύνολο ψηφίσματος τροπολογία 1 Περ κατά αποχέ εγκρίνεται σύνολο ψηφίσματος ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκτε Αρβαμά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έλεγχο τη Αλία. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματο μοναστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται τώρα έκθεση Αρβαμά για την Ευρωπαϊκή Αρχή την Ασφάλεια των Τροφίμων. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο ψήφισμα έχουμε τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έγινε δεκτή τροπολογία. Τώρα το σύνολο ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην εξαρβαμά για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Απόφαση για την απαλλαγή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Θέλετε να ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έγινε δεκτή. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Έκθεση Αρβαμά τώρα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Αρβαμά για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται σύνολο ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα έχουν τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται Έκθεση Αρβαμά για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία. Απόφαση την απαλλαγή ψηφιπέρ. Κατά. Ποχέ. Εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματο. μονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Απόφαση για την απαλλαγή ψηφιπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος, μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκθεσαρβάμα Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος, μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Έκτε αρβάμα για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση για την αυλαγή υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματο. Μάλλον έχουμε την τροπολογία καταρχά 1. ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ. Ελέγχουμε παρακαλώ την τροπολογία 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η ένα και πηγαίνουμε στο σύνολο του ψηφίσματο ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Σαρβαμά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Απόφαση να βλαγεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται εξαρβαμά για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής εκπαίδευση. Απόφαση για την απαλλαγή κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. Η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκταση αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων τη μεγάλη κλίμακα στον χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ψήφι υπέρ τη απαλλαγή. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση τώρα για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται έκθεση Αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος μοναστική εκκλησία για την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Σαρβαμά για τον Οργανισμό Εφοδιασμού τη Ευρατόμ. Ψηφίζουμε την απαλλαγή υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματο μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται εξαρβαμά για το Ευρωπαϊκό Έδραμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωση και Εργασία. Απόφαση την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται από σύνολο ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται εξαρβαμά για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μάλλον η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστική Συνεργασία περκατά αποχέ για την απαλλαγή. Ονομαστική κλίση για το ψήφισμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στην έκθεση Αρβάμα για τον οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνεργασία των Μετσαπιπολιτών. Περκατά αποχέ για την απαλλαγή. Ψήφισμα. Αρχικό κείμενο τη 10. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο του ψηφίσματος μας κλείσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκτε αρβαμά για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε την απαλλαγή υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση στο σύνολο του ψηφίσματο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Έκθεση Αρβαμά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φυλακή και Ακτοφυλακή. Ε, το ψήφισμα, μάλλον απόψη θα κατά αποχέ εγκρίνεται. Στο ψήφισμα έχουμε τροπολογία ένα ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται το σύνολο του ψήφισματο μονομαστική κλίση. έρχεται ψηφοφορία. Ψηφισάτε όλοι πέρα. Εγκρίνεται τώρα εκδαβάμα για τον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS. Ψηφίζουμε την απαλλαγή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος μας στην κλεισά και ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε κάποιες εκθεσούλες της κυρίας Ντλαμπάγιοβα. Κοινή επιχείρηση βιομηχανικών δύο πρώτων καταρχάς Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, η έκθεση Λαμπάγιοβα για την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Ψηφίζουμε την απαλλαγή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο ψήφισμα μοναστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την έκθεση Λαμπάιοβα για, για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία. Απόφαση την απαλλαγή ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται τώρα έκθεση Τλαμπάγιοβα για την κοινή επιχείρηση Κυψέλε Καυσίμου και Υδρογόνο, απόφαση για την απαλλαγή. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σύνολο ψηφίσματος. Ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται έκθεση Τλαμπάγιοβα για την κοινή επιχείρηση πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2. Απόφαση την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα τη Λαμπάγιοβα για το ΙΤΕΡ και ανάπτυξη κοινή επιχείρηση πυρηνική σύνδεξη για την απαλλαγή ψηφισμού. Πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απόφαση το σύνολο της ψηφίσματος μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα έκθεση Λαμπάγιοβα για την κοινή επιχείρηση Σέζαρ. Ψηφίζουμε την απαλλαγή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και τώρα τελευταία